Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξέρω ότι είχαμε ε, Έχουμε τη συνέχεια μιας πολύ ενδιαφέρουσας συνεδρίασης με τον πρόεδρο ε, Ρούμπικ ε, για την ε, έκθεση για την εθνική εφαρμογή. Είναι η πρώτη τέτοια έκθεση που παρουσιάζουμε. Ακούσαμε πάρα πολλά στοιχεία και εμπειρίες για το θέμα αυτό και μας τιμά αυτή η συνεργασία. Τώρα θα συνεχίσω στα Ιταλικά, αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα απλώς να πω ευχαριστώ στον κύριο Ρούμπικ που είναι παρόν και αντικαθιστά τον πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε τον κύριο Μπούζεκ, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρεθεί διότι είναι στην Αυστρία. Ε, now I, ε, we begin our joint... Και ξεκινούμε λοιπόν την κοινή μας συνεδρίαση. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Ε, ελπίζω να μην είναι και η τελευταία. Θα περάσω και στα Ιταλικά, είναι καλύτερα για μένα και για σας. Καταρχά πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, ω τροποποιήθηκε. Από ό,τι βλέπω, ναι, υπάρχει διερμηνία σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά. Βεβαίως, ε, η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά μέσω web streaming δεν είμαστε πολλοί, αλλά νομίζω ότι υπάρχει εκπροσώπηση από όλες τις πολιτικές ομάδες, επομένως είναι καλή εκπροσώπηση και ε, είναι η ώρα αυτή τη κοινή πρωτοβουλία. Έχουμε λοιπόν σήμερα αυτή την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ήτρε για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να σα ζητήσω λίγο ησυχία, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη. Λίγο ησυχία. Ευχαριστώ. Για να γίνει λοιπόν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο κοινή έκθεση, ε, το οποίο επιθυμούσαμε διακαώς, ε, μια συνεκτική πολιτική για την πολιτιστικέ και δημιουργικέ βιομηχανίε ευρωπαϊκή Ένωση. Να συγχαρώ ευθύ εξ αρχή του ε, δύο εισηγητές, τους κυρίους Έλλερ και Μόργανο, για την αγαστή συνεργασία και για τα όσα έκαναν ε, ήταν πολύ έντονε εργασίε και είναι και η πρώτη φορά που η Επιτροπή Ήτρε και η Επιτροπή Πολιτισμού συνεργάζονται για ένα κείμενο το οποίο έχει προκύψει από κοινή ε, διάθεση και κοινό ενδιαφέρον για την ε, δημιουργική και ε, πολιτιστική βιομηχανία, μετά την Πράσινη Βίβλο, μετά από την πρώτη έκθεση που έκανε η κυρία Σάντσε Σμιθ ε, στην προηγούμενη θητεία και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε εκ νέου μια στρατηγική η οποία κατά την άποψή μα έχει ε, ελάχιστη εφαρμογή, ελάχιστη παρακολούθηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς θεωρούμε ότι ο τομέα αυτό στην Ευρώπη είναι ένα από του πιο πολλά υποσχόμενου τομεί Αναφερόμαστε πλέον σε ένα 5% του ΑΕΠ και περίπου 8.000 ε, θέσεις ε, είναι και ένας τομέας ο οποίος ε, στη διάρκεια της κρίσης πήγε ενάντια στο ρεύμα, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε και σε μια δουλειά ε, αριστείας και από πλευράς κατάρτισης και πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τομέα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και ε, προσδίδει αξία σε αυτή την πολιτιστική ποικιλομορφία και στην βιομηχανική ποικιλομορφία που είναι το πιο σημαντικό μας χαρακτηριστικό. Και πιστεύω ότι αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ε, είμαστε τόσο ικανοποιημένοι για την έναρξη αυτής της συνάντησης και μπορούμε να συνεργαστούμε για μια έκθεση η οποία λογικά θα δώσει και μια πολύ σημαντική όθηση στις προτεραιότητες του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δώσω τώρα το λόγο για να απευθύνει χαιρετισμό και να του πω και πάλι ε, καλώς ορίσατε στον πρόεδρο, συμπρόεδρο σε αυτή την περίπτωση, στον κύριο Ρούμπικ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι Κώστα, η Συνάδελφο και συμπροέδρο ε, φέρει μεγάλη ευθύνη από κοινού με συναδέλφου από την Επιτροπή Κουλτ και Ήτρε και χαίρομαι που πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση που λαμβάνει η χώρα σε οριζόντιο επίπεδο και για το γεγονό ότι και οι δύο επιτροπέ επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο αυτό θέμα από τον βιομηχανικό κλάδο και θα εξετάσουμε από εκείνο το θέμα αυτό. Η πολιτισμική βιομηχανία θα αποτελέσει ένα άλλο ένα και πιο σημαντικό θέμα γιατί ζούμε μια επανάσταση σε μια εποχή επαναστατική. από τον ε, πραγματικό κόσμο περνάμε και αντικατοπτριζόμεθα στον ψηφιακό κόσμο και στον ψηφιακό κόσμο περιλαμβάνονται και πολλές καινούργιες ευκαιρίες, πολλές καινούργιες δυνατότητες, κωδικοποίηση και άλλες νέες μορφές επικοινωνίας, social media. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία καλούν τους νέους μας να τα χρησιμοποιήσουν και είναι νομίζω σημαντική πρόκληση αυτή. Ξέρουμε ότι 12 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ε, μπορούν να δημιουργηθούν, οι οποίες θα σημαίνουν και σημαντικά έσοδα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και την συνολική, το συνολικό αντίκτυπο της βιομηχανία ε, πολιτισμού και οι εμπορικές συμφωνίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο σημείο αυτό σε ό,τι αφορά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την πολιτισμική βιομηχανία. Και βλέπουμε επίσης ότι η πολιτισμική βιομηχανία και στο μέλλον θα συνεχίσει να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, γιατί νομίζω ότι είναι στην αιχμή του τόρτος η Ευρώπη. Η Ευρώπη του 21ου αιώνα θα είναι διαφορετική και θα διαμορφωθεί και θα εξελιχθεί σημαντικά. Προσβλέπω λοιπόν στη σημερινή συνάντηση, γιατί εδώ πέρα πιστεύω ότι υπάρχουν ευκαιρίε για του πολίτε μα ό,τι αφορά την υποθέτηση και την ε, θέση τη Ευρώπη στον κόσμο. Δηλαδή, δεν θέλουμε να καταρρεύσει η Ευρώπη, θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη και αυτό είναι το μέλλον μα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο Ρούμπιχ. Μπορούμε να δώσουμε απευθεία το λόγο στους δύο συνεισηγητές και να προσθέσω ότι εάν δούμε τα άτομα που ασχολούνται με την δημιουργική ε, βιομηχανία ε, και την πολιτιστική βιομηχανία είναι ε, διπλάσια από την βιομηχανία και σχεδόν τριπλάσια από τη χημική βιομηχανία θα μπορέσουν ίσως να καταλάβουν και οι πιο δύσπιστοι πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση. Έχουμε μια πιο αριζόντια εργασία όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, εμένα μου αρέσει να κάνω διάκριση ε, μεταξύ των αρμοδιοτήτων και να έχουμε μια πιο οριζόντια στρατηγική και δεύτερον, διότι εδώ θεωρώ ότι μας ενδιαφέρει να συνομιλήσουμε και ε, όσον αφορά τις βασικές προκλήσεις και τις τεχνολογίες αλλά και τις δεξιότητες που είναι ένα επόμενο πακέτο που έχουμε και το στρατηγικό ταμείο ε, για τη επενδύσεων που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Έλλερ. E για πέντε λεπτά και μετά στο Λίτζι Μόργανο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Ρούμπιχ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, και αυτή δεν είναι η συνήθις ευρωπαϊκή ευγένεια. Θέλω να ευχαριστήσω πολλούς ανθρώπους. Αυτή η κοινή προσπάθεια έδειξε ευθύ εξ αρχή ότι εργαζόμαστε με ένα κείμενο. Ε, συνήθως έχουμε μια διαδικασία του άρθρου 50 και ξεκινάει η μάχη. Ευθύ εξ αρχή, εμεί όμω είχαμε δύο γραμματείε με κάποιε κατευθυντήριε από γραμμέ από του ηγητέ και εργαζόμασταν για ένα κοινό κείμενο και αυτό ήταν ένα πολύ θετικό τρόπο εργασία και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Να ευχαριστήσω και τους δύο προέδρους, διότι υπήρξαν φόβοι στην αρχή ε, πώς θα ε, επηρεάζει η έκθεση αυτή τη υποχρεώσεις τη μια επιτροπή και τη άλλη, νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Να ευχαριστήσω πολλέ ε, κυρίε γιατί μπορεί να αναφερθώ στην ε, ομάδα τη Δημιουργική Βιομηχανία και το, οι δύο εισηγητέ ε, είναι ε, ταπεινοί υπηρέτε ανδρών και γυναικών. Να ευχαριστήσω την κυρία Τρούπελ, την κυρία Φερχάιν, την Περβάν Σπερέ και πολλέ άλλου συναδέλφου οι οποίοι βοήθησαν να προωθήσουμε την ιδέα ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε από κοινού και να αναφερθούν ε, στη σημασία της δημιουργικής βιομηχανίας, να έχουμε περισσότερα κονδύλια, μεγαλύτερη συνοχή και περισσότερες συνέργειες μεταξύ της χρηματοδότησης και των χρηματοοικονομικών μέσων. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε μεταξύ των στοιχείων που σας παρουσιάζω τώρα, διότι χρειάστηκε κάπου λίγο να γίνει ένας διαχωρισμός για την προοπτική της Επιτροπής Βιομηχανίας, αλλά είναι κοινή έκθεση και συμμεριζόμαστε πλήρως τις απόψεις της Επιτροπής Πολιτισμού και αντιστρόφους, αλλά είμαστε δύο εισηγητές και μπορεί εγώ να ε, αναφέρομαι περισσότερο στα θέματα της βιομηχανίας και ο Λουίτζι έχει περισσότερο τις απόψεις της Επιτροπής Πολιτισμού, αλλά είναι κοινή έκθεση. Τα στοιχεία που είναι σημαντικά γιατί δεν έχει γίνει αντιληφθού μέχρι τώρα ε, σε τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν το έχουν αναγκαλίσει και τα κράτη-μέλη, είναι το γεγονός ότι η δημιουργική βιομηχανία στην Ευρώπη, και αυτό πρέπει να γραφτεί στον εγκέφαλό μας, παρέχει πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Είναι ε, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, του, εργατικού δυναμικού, 550 δις προσθήκη στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ και συνεισφέρει περίπου στο 5% του συνολικού ΑΕΠ και είναι περίπου το 5% των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 2,5 φορέ φορές περισσότερα άτομα από ό,τι στην αυτοκινητοβιομηχανία και ε, τέσσερι 4 φορές περισσότερο από τη χημική βιομηχανία. Και αν δείτε συγκεκριμένους τομείς στον ορίζοντα 2020 που σχετίζονται με πιο μικρού κλάδου, έχουμε διπλάσια ή τριπλάσια χρηματοδότηση για έρευνα. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι λίγο ε, πολύ δείχνει πόσες ελλείψεις υπάρχουν ε, στα θέματα και τα προγράμματα της δημιουργικότητας. Νομίζω ότι πέραν όλων αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν έχει μια συνεκτική βιομηχανική πολιτική για αυτό τον τόσο σημαντικό τομέα και είναι ίσως και ο τελευταίο τομέας που θα μπορούσαμε να ασπαστούμε στον τομέα αυτό. Αλλά αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ασχολείται με διάφορα θέματα, ασχολείται με ψηφιοποίηση, πνευματικά δικαιώματα, πολιτιστική κληρονομιά, χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, χρηματοδότηση για πολιτιστικέ δραστηριότητε που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αλλά ουσιαστικά δημιουργούμε ένα πλαίσιο νομοθεσία, υπάρχουν ρυθμιστικέ προσπάθειε, δεν έχουμε όμω επικεντρωθεί στον κλάδο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό, να γίνει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποια από τα στοιχεία που παρουσιάζουμε στην έκθεση βασίζονται σε μια μελέτη που θα δημοσιεύσει μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε λίγες ημέρες. Υπήρξε στενή συνεργασία λοιπόν με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση και τις υπηρεσίες μας, αλλά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερη δραστηριότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός της έκθεσης είναι να εντοπίσουμε τα βασικά στοιχεία που ενδιαφέρουν όλους. Ε, ο πολιτιστικό τομέα στην Ευρώπη μπορεί να είναι διαφοροποιημένος αλλά όλοι έχουν τις ίδιε ανησυχίε, όπως για παράδειγμα πρόσβαση στη χρηματοδότηση, προώθηση νέων ταλέντων και ανάπτυξη δεξιοτήτων και καινοτομία. Επιπλέον, στον 21ο αιώνα η μετάβαση η οικονομία σημαίνει ότι έχουμε αντικατάσταση ε, των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής και ο αναγνωρισμένος ορισμός του, είναι, του τι είναι πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία μπορεί να είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που ο κλάδος δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί ως ένας τομέας ο οποίος είναι συγκρίσιμος με άλλους κλάδους όπως για παράδειγμα την αυτοκινητοβιομηχανία. Το πρώτο μας βήμα κατά την εκπόνηση της ε, έκθεσης ήταν να προτείνουμε ε, τον εξή ορισμό ο οποίος θα αποτελέσει βάση για τις μελλοντικέ δραστηριότητες ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Καθυστερήσαμε λίγο για να μπορέσουμε να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά. Ο ορισμός θα είναι Πολιτιστικέ και δημιουργικέ βιομηχανίε είναι αυτέ οι οποίε βασίζονται σε πολιτιστικέ αξίε, ατομική δημιουργικότητα, δυνατότητα δημιουργία θέσεων εργασία μέσω αξιοποίηση τη πνευματική ιδιοκτησία και περιλαμβάνουν τομεί που βασίζονται σε πολιτιστική και δημιουργική συνεισφορά, αρχιτεκτονικά έργα, βιβλιοθήκε, καλλιτεχνικά έργα, ε, λογισμικό που περιλαμβάνει και video game και οπτικοακουστικά μέσα, ε, μόδα, φεστιβάλ, μουσική, ε, τέχνες, δημοσιεύσεις, ε, ραδιόφωνο και ε, visual arts. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά γιατί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται ε, σημαίνει ότι οι αρμόδιοι φορές ελάχιστα αναγνωρίζουν τις πλήρες δυνατότητες του συγκεκριμένου κλάδου. Όπως σας είπα αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι χρειαζόμαστε πολιτικές κομμένες και ραμμένες στα μέτρα αυτών των, κλάδων και αυτό σημαίνει ε, λύσεις ε, στον τομέα της χρηματοδότησης ε, κυρίως πρέπει να ευθυγραμμώσουμε τα προγράμματα χρηματοδότησης, να είναι προτεραιότητα στον ορίζοντα 2020, ιδιαιτέρως πρέπει να υπάρχει πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και να εκμεταλλευτούμε πιθανές ενέργειες που υπάρχουν μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών και νέων προγραμμάτων. Οι ε, περιφέρειες είναι πολύ καλέ στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δομών. Μήπως μπορείτε να ολοκληρώσετε, γιατί καθυστερείτε, διακόπτη Πρόεδρο. Ναι, ναι, τελειώνω. Τι πρόθεση έχουμε λοιπόν. Πρέπει ουσιαστικά να ορίσουμε τον τομέα και πρέπει να την χάνει ισότιμη μεταχείριση με άλλου τομεί στην Ευρώπη. Πρέπει να ευθαγραμμίσουμε τα προγράμματα. Θέλουμε να έχουμε περισσότερες κοινέ ε, προσκλήσεις ε, προσφορών και θέλουμε να ενισχύσουμε την ιδέα ότι ακόμα και θέματα ε, που αφορούν την εκπαίδευση των νέων μπορούν να αφορούν και το συγκεκριμένο κλάδο. Και επίση πρέπει να αναφερθούμε πολύ στην εκβιομηχάνηση τη Ευρώπη. Η δημιουργική βιομηχανία μπορεί να είναι ένα από του βασικού κλάδου που μπορεί να βοηθήσει στην εκβιομηχάνηση τη Ευρώπη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να γίνει αντιληπτό και είναι ο στόχο μα πολύ πέρα τη έκθεση. Δεν είναι ο... το τέλο, είναι η αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μόργανο έχει το λόγο. Πέντε λεπτά το πολύ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους εγκαρδίους όπως και ο κύριος Έλερ και να ευχαριστήσω και τον ίδιο τον κύριο Έλερ. Τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία χρησιμεύσαν σαν σημείο κίνησης αυτής της πρωτοβουλίας. Ένα άλλο σημείο ήταν το επίπεδο ορισμού, τον οποίο θελήσαμε όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται για να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα των χρηματοδοτήσεων. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες μικρές υπογραμμίσεις λαμβάνοντας απλά τις δυνατότητες σε επίπεδο χρόνου τις οποίες έχουμε. Νομίζω ότι έχει σημασία να υπογραμμίσουμε τον διοικό χαρακτήρα της ε, ε, ρητορική μας, αν θέλετε. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη σχέση τέχνης, πολιτισμού, οικονομίας και τεχνολογίας. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την ανάγκη ε, προστασίας της γλωσσικής ποικιλία της Ευρώπης, της ηλικής αλλά και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, να δούμε τι ε, γίνεται με τις καινοτομίες ε, σε ορισμένους τομείς όπως το λιανικό εμπόριο, ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα έλεγα δεν αποκρύβεται σε σχέση με την πολιτιστική ευρωπαϊκή διπλωματία και υπάρχει επίσης και η ανάγκη να θεωρήσουμε με κάποιο τρόπο ε, να αναζητήσουμε με κάποιο τρόπο την απάντηση στην ε, κρίση στον τομέα της απασχόλησης. Σε αυτήν την οικονομική δραστηριότητα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα, εργάζονται νέοι. Η πλειοψηφία αυτών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, των οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι μικροεπιχειρήσεις με κάτω από 9 εργαζομένους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν το 90% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Νομίζω λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό να υπογραμμίσουμε ότι μετά την οικονομική κρίση του 2008 ο τομέας αυτός ήταν ο πλέον ανθεκτικό. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι παρουσίες ε, δραστηριότητας οικονομικής οι εταιρείε αυτές που δύσκολα μετακινούνται σε άλλες χώρες. Έχει σημασία λοιπόν αυτό τώρα για την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά μένει να γίνουν. Πάντως το θέμα είναι τα παιδιά να αποκτούν ήδη από μικρή ηλικία τις ε, ικανότητες που απαιτούνται στο σχολείο. Τίθεται θέμα εδώ ε, της διδακτικής ύλης, θα πρέπει οι προτάσεις αυτές να ε, υποστηριχθούν. Η επιλογή της παρέμβασης στην τυπολογία αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων, των ε, δραστηριοτήτων λοιπόν στον τομέα του πολιτισμού, είναι κάτι το απαραίτητο. Πρέπει να έχουμε λοιπόν σωστά προπαρασκευασμένους ανθρώπινους πόρους οι οποίοι να μπορέσουν να χρησιμεύσουν στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας. Ε, για τα υπόλοιπα θα συμφωνήσω με τον κύριο Έλλερ ότι θα πρέπει να διευρύνουμε ορισμένους τομείς και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και στην τεχνική και ε, ε, δευτερα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όλα αυτά προσθέτουν νομίζω σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το θέμα είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στην ευρύτερη δυνατή πολιτική συνένεση, να στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πιο ξεκάθαρη λύση, ότι δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι δεν μπορούμε να αναβάλουμε πλέον μία πολιτική στον τομέα αυτό η οποία να είναι συνεκτική και στις δημιουργικές αυτές οικονομικές δραστηριότητες. Όλα αυτά τα έχει ήδη υπογραμμίσει ο κύριος Σέλερ και άπτονται του θέματος της χρηματοδότησης, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, κατανοώντας σωστά το στρατηγικό ταμείο, το ΕΦΣΥ, και να δούμε επίσης τι γίνεται και με τον μηχανισμό εγγυήσεων δημιουργικού η Ευρώπη, που θα μπορούσε και μέσω του ΕΦΣΥ να λειτουργήσει καλύτερα. Πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις, πρέπει να καταπολεμήσουμε την παραποίηση των προϊόντων, πρέπει να προστατεύσουμε την πνευματική ιδιοκτησία, να σημειώσω προς τους συναδέλφους ότι έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα που λύθηκαν ε, στις μεταφράσεις προς τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά της πρότασης. Τώρα πλέον οι γλωσσικές αυτές, ε, ε, οι εκθέσεις σε επίπεδο γλωσσικό είναι σωστές και στις γλώσσες αυτές. 6 ε, Σεπτεμβρίου μία κατάθεση των τροπολογιών, το λέω αυτό για να μην ξεχαστεί. Να πω επίσης ότι σε μία έκθεση για... με το χώρο και το μέγεθος που μπορεί να έχει, δεν μπορούμε να βάλουμε τα πάντα, αλλά με τον συνάδελφο Έκλερ θα καταθέσουμε από κοινού κάποιες κοινέ τροπολογίες για να συμπληρώσουμε το πλαίσιο που επιθυμούμε. Σας ευχαριστώ. Φαίνεται ότι έγινε συνολική προσπάθεια, λέει η πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω τώρα τον λόγο για τον πρώτο γύρο στους σκιώδεις εισηγητές. Και στον δεύτερο γύρο θα, προεδρεύσει ο κύριος Ρούμπικ, θα ομιλήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Μπόγκταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους συζητητές. Η έκθεση αυτή είναι εξαιρετική. Τα πιο σημαντικά ζητήματα αποτυπώνονται στην έκθεση. Στη δεκαετία του 90 ήδη σημειώθηκαν ε, μεγάλες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Πολιτισμική και Δημιουργική Βιομηχανία. Αυτό δημιούργησε θέσει εργασία και είχε σημαντικό μερίδιο στο ΑΕΠ. Χρειαζόμαστε στρατηγικέ επενδύσει λοιπόν υπέρ τη ε, πολιτισμική πολυμορφία, τη κοινωνική συνοχή, των θέσεων απασχόληση και τη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μια ευρεία πολιτισμική προσφορά ψηφιακού περιεχομένου. Αυτό θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε μηνύματα βάσει των ευρωπαϊκών αξιών. Η δημιουργική βιομηχανία προωθεί και την ε, καινοτομία, την τεχνολογική καινοτομία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και θα πρέπει να προωθήσουμε την κινητικότητα μεταξύ των καλλιτεχνών γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον οικονομικό κλάδο που ασχολείται με τα πολιτισμικά, προκειμένου να περάσουν από το περιφερειακό στο εθνικό επίπεδο. Για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, χρειάζεται βιώσιμε εταιρικέ σχέσει μεταξύ των ε, απασχολούμενων στον κλάδο βάσει τακτικών διαβουλεύσεων. Πρέπει να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στον κλάδο αυτό και να φροντίσουμε να τα εμπόδια τα οποία εμποδίζουν την κινητικότητα. Θα πρέπει να αξιοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό προϋποθέτει αρρωγή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ το CCI. Μα μέσω και μακροπρόθεσμα αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένε αλλαγέ. Σε ό,τι αφορά την φορολογία, για παράδειγμα, θα πρέπει να προσαρμοστεί. Και αυτό το αναφέρω ήδη παραδείγματο. η ΕΤΕΠ και η σχετική χρηματοδότηση ή η χρηματοδότηση μέχρι του ΕΦΣΙ, άλλη μια πηγή. Αν θέλουμε η δημιουργική βιομηχανία να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της ως προς την δημιουργικότητά της, θα πρέπει να δώσουμε σωστή πρόσβαση στη χρηματοδότηση και το σύστημα το φορολογικό θα πρέπει να α, ικανοποιήσει τις ανάγκες του συστήματος. Θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε το πλήρες δυναμικό του CCI. Αυτό θα σήμαινε και σωστή εκπαίδευση και κατάσταση στα σχολεία. Ευχαριστώ και γιατί σέβεστε το χρόνο. Ο συνάδελφος ε, Χωσέ Μπρανκο Λόπες από την Επιτροπή Ήτρε τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς ε, για το έργο των ε, συνεισηγητών πολύ εύστοχοι στις παρατηρήσεις τους για τα προβλήματα χρηματοδότησης της πολιτιστικής και βιομηχανίας και δημιουργικής βιομηχανίας και όσον αφορά την αναγνώριση και την ε, κατάρτιση ε, στον τομέα αυτό από τα σπάργανα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η βάση για τα όσα πρέπει να ε, κάνουμε στη συνέχεια. Είναι περίπλοκο να καθορίσουμε το βάσορος της πολιτισμικής και δημιουργικής βιομηχανίας και εκφύσεως και λόγω έλλειψης κοινών ορισμών και πλήρων στατιστικών στοιχείων. Παρόλα αυτά, Πέραν ε, του ποσοστού του ΑΕΠ, όπως μας είπε και η Πρόεδρος, ε, η δημιουργική και η πολιτιστική βιομηχανία έχουν αποδείξει ότι αντέχουν ε, στην κρίση και μπορούν να συνεχίσουν να δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση όταν άλλοι τομείς ε, την καταστρέφουν. Η πολιτιστική βιομηχανία κυρίως ε, προσδίδουν αξία στην επανάσταση που βιώνουμε. Είναι πηγή δημιουργικότητας, πηγή καινοτομίας, διαφοροποίησης και αποτελούν τη βάση, ε, βάση της ε, επιθυμητής ψηφιακής βιομηχανίας, το περιεχόμενο δηλαδή. Ε, η επανάσταση η οποία έρχεται πρέπει να γίνει ε, με ενίσχυση της προστασίας, καταπολέμηση της παρατποίησης και της πειρατείας, καταπολέμηση επίσης ε, της στέρηση των δικαιωμάτων των δημιουργούν λόγω της ψευδούς έλλειψης ευθύνης που υπάρχουν για το περιεχόμενο που διαδίδεται ψηφιακά κλάδος θα ενισχυθεί αν μπορέσουμε να προστατεύσουμε το βασικό του κεφάλαιο. Και το βασικό κεφάλαιο δεν είναι άλλο ε, παρά η πνευματική ιδιοκτησία. Και τέλος, και με αυτό ολοκληρώνω, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να σκεφτούμε και να ενισχύσουμε στην έκθεση την κοινωνικο-εργατική σχέση της ε, πολιτιστικής βιομηχανίας η έλλειψη ενός συγκεκριμένου εργατικού πλαισίου που να αναφέρεται στις ιδιωτερότητες του τομέα, η ανάγκη να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για τους εργαζομένους και να λάβουμε υπόψη τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που υπάρχουν και σε θέματα κινητικότητας. Είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε ένα καρποφόρο διάλογο και θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Μακλάκινγκ. Δεν σας είδα, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και θα πρέπει να τονίσουμε και να δώσουμε έμφαση στο πόσο σημαντικές είναι αυτές, ε, αυτή η κλάδη για μας. Και είναι καλό λοιπόν που συνεργάζονται και οι επιτροπές. Η σημασία λοιπόν των ζητημάτων αυτών για, το, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ σημαντική. Πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια πρώτη πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων. Θα πρέπει να σκεφτούμε όμως το πώς θα επιδείξουμε και θετικό χαρακτήρα και αισιόδοξο χαρακτήρα προκειμένου να βοηθήσουμε τους κλάδους αυτούς να αναπτυχθούν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε σήμερα για να είμαστε πρωταθλητέ ε, στο θέμα αυτό και να είμαστε και χρήσιμοι και ωφέλιμοι στι προτάσει, μα χωρί να υπονομεύσουμε τα επιχειρηματικά μουλά τα οποία ήδη ε, αποφέρουν καρπού και λειτουργούν αποδοτικά σε κάποια σημεία και να μην ε, παρεμποδίσουμε τις ανάγκες του κλάδου. Θα ήθελα να επικεντρωθώ λοιπόν στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησίας, των διεθνών δικαιωμάτων και να δούμε πώ μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η αξία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας αυτό και να υπάρχουν και εργαλεία για να προστατεύσουν τα πνευματικά αυτά δικαιώματα. Νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως την καταπολέμηση του παράνομου κατεβάσματος από το διαδίκτυο και το τι ζημία προκαλεί αυτό στην, ε, στο κλάδο. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους ε, παραγωγούς μου και τους καλλιτέχνες. Έχω και κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των καλλιτεχνών. Και πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει σωστή αποζημίωσή τους για να αξιολογείται σωστά και η δουλειά τους και τα προϊόντα τους και η πολιτισμική αξία των προϊόντων τους και ιδιαίτερως δεδομένης και της νέας τεχνολογίας, βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα streaming, για παράδειγμα, και άλλες πολλές τεχνολογικές δυνατότητες που αποτελούν τεράστια πρόκληση για τους ε, καλλιτέχνες και τους δημιουργούς. Δεν πιστεύω ότι στην παρούσα φάση πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ε, νομικού πλαισίου, να σεβαστούμε την ελευθερία του ατόμου και να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την διαφάνεια. Γιατί αυτό μπορούμε να το κάνουμε για να βοηθήσουμε τον καλλιτέχνη και τον δημιουργό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ε, βαρύς μηχανισμός, ε, νομοθεσίας. Ενδεχομένω να υπάρχουν άλλοι πιο ελαφροί μηχανισμοί οι οποίοι να βοηθούν καλύτερα, για παράδειγμα, στη διαπραγμάτευση συμβάσεων να ενημερώνονται σωστά οι δημιουργοί για τι ε, συμβατικέ του ε, ελευθερίε, τα συμβατικά του δικαιώματα. Πολλά λοιπόν ε, μπορούμε να συζητήσουμε και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι γίνεται και με την οδηγία για τι οπτοακουστικέ υπηρεσίε, για να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι συναντιόμαστε σήμερα και είναι σημαντικό να συζητήσουμε συνολικά το πώ ε, θα βελτιώσουμε την κατάσταση για όλον τον πλάτο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο, Και τώρα από την ε, Επιτροπή Ήτρε, η συνάδελφο Αντζέλη Καμινέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και του δύο εισηγητές ε, και τον κύριο Μοργάνο και τον κύριο Έλλερ από την Ήτρη για την καλή δουλειά που έχουν κάνει και χαίρομαι ιδιαίτερω που κάνουμε τη συζήτηση αυτή εδώ σήμερα και συνεργαζόμαστε για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Δυστυχώ, ο ε, πολιτισμικό κλάδο αυτό και ο κλάδο των δημιουργών δεν είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων τη Επιτροπή και τη ΙΤΡΕ. Και παρά το γεγονό ότι ξέρουμε τι σημαίνουν για τι θέσει απασχόληση. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεση των δύο συνεισηγητών και προσβλέπω στην ε, κατάθεση και δικών μου προτάσεων. Τα πιο πολλά σημαντικά ζητήματα για τον πολιτισμικό κλάδο είναι η δυσκολία του ορισμού μεταξύ των κρατών μελών, των επαγγελμάτων, θέματα συγκρίσιμότητας, θέματα αμοιβαιότητας, η πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Ωστόσο, πιστεύω ότι κάτι άλλο θα πρέπει να τονίσουμε, γιατί είναι πολύ επικαιρή αυτή η έκθεση οι τεχνολογίες αυτές περνάνε από φάση τεράστιας αλλαγής ε, στην τεχνολογική εποχή και θα πρέπει να δράξουμε πλήρως τα ωφέλη που προσφέρει η ψηφιοποίηση, γιατί αυτό ουσιαστικά επεκτείνεται και σε όλους τους άλλους οικονομικούς κλάδους, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τεχνολογίες επικοινωνίας, αποτελούν κινητήριες μηχανές για την οικονομία στην ψηφιακή εποχή και έτσι συμβάλλουν στην καινοτομία. Τα CCI λοιπόν αποτελούν σημείο κίνησης για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και για νέε καινοτομίε. Είναι σημαντικό να λεφθούν πιο πολύ υπόψη λοιπόν ακόμα και να καθιστούν προτεραιότητα στην τεπάρτιση νομοθεσία στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να δούμε και τις πολιτικές πρωτοβουλίε, όπως είναι η υπηρεσία για τα όπτιο ακουστικά, οι πολιτικέ για τον αποκλεισμό τα θέματα copyright, όλα αυτά πρέπει να λεφτούν υπόψη για να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα και των πατών και των δημιουργών. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει ένα εύρυθμα λειτουργών σύστημα στην Ευρώπη, όπω αναφέρεται και στην έκθεση, με όλου του εμπλεκόμενου φορεί για να υπάρχει σωστή πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να υπάρχουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ε, εταιρικέ σχέσει. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται σε πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ο λόγος τώρα στο κύριο Μυρτσία Διακόνο από την Επιτροπή Πολιτισμού από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Έλερ, γιατί ο κύριος, ο κύριος Μόργαν είναι φίλος μου και δεν χρειάζεται να τον ευχαριστώ και δημοσίως. Του τα έχω πει διαζώσεις. Όταν ε, ε, ήμουν εγώ αρμόδιος για την ε, προσέγγιση για την πολιτισμική κληρονομιά στην Επιτροπή μας, ε, είδαμε τι γίνεται με τον προϋπολογισμό των κρατών μελών, προϋπολογισμό για τον πολιτισμό, για την πολιτισμική κληρονομιά κλπ. Και τότε είχα κρατήσει κάποια στοιχεία, κάποιες συγκρίσεις για τη σχέση μεταξύ του προϋπολογισμού που υπάρχει και τις ανάγκες του τομέα. Ε, τώρα διάβασα την έκθεση και βλέπω τα πραγματικά στοιχεία της ε, οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Η συνεισφορά του πολιτισμικού τομέα είναι τεράστια σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουμε στον προϋπολογισμό ε, σε εθνικό επίπεδο για τον πολιτισμό. Κάποια από τα κράτη-μέλη μας συνεισφέρουμε γελίο ε, ποσά στο ε, πολιτισμό. Παραδείγματο χάρη, η χώρα, μου δίνει 0,03% του προπολογισμού της ε, σε πολιτισμό. Για τα στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μία πρόταση στους συνεισηγητές. Φυσικά θα μπορούσα να υποβάλω και σχετική τροπολογία. Σας προτρέπω λοιπόν να ζητήσετε, να προτείνετε στα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν ε, την ε, ε, αντίληψη που έχουν για το θέμα και να αλλάξουν και αντιστοίχω τον προπολογισμό. Να αλλάξει δηλαδή η αντιμετώπιση προς τον πολιτισμό. Διότι προς το παρόν λέμε ότι η χρηματοδότηση είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προκύπτει και από το εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ τον κύριο Διακόνου. Και τώρα ο λόγος στην Μαρτίνα Μίκελς από την ΚΟΕ, από την Επιτροπή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους εισηγητές για την ε, πάρα πολύ σημαντική για μας ε, έκθεση. Τέτοια θετικό... Οι είναι οι εντυπώσεις ε, και συμφωνούμε ιδιαίτερως με τη διεύρυνση του όρου της ε, οικονομίας, ε, πολιτισμού και δημιουργικότητας για να συμπεριληφθούν νέα στοιχεία. Ωστόσο, είναι όλα αυτά πολιτισμικά προϊόντα. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν και οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με, την, ε, με τον πολιτισμό όπως είναι η διακίνηση, η διαμεσολάβηση έργων τέχνης, γιατί είναι και αυτά πάρα πολύ χρήσιμα. Το έχετε λάβει αυτό υπόψη. Εγώ θα το υποστήριζα. Και μία παρατήρηση για τα χρηματοοικονομικά μέσα και την χρηματοδότηση. Έγινε ήδη μία σύνδεση στο, με το ΕΦΣΥ. Από την άλλη βέβαια, δυστυχώς στην παρούσα φάση ως το Μάιο του 2016 αναγκαστικά πρέπει να σκίσουμε και ε, κριτική ε, για το ΕΦΣΙ. Γιατί κανένα από τα project δεν, ε, το CCI δεν χρηματοδοτήθηκε από το ΕΦΣΙ. Και τώρα ό,τι αφορά τα 121 εκατομμύρια από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά πόσον θα υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα το δούμε. Θα πρέπει να γίνει μια εις βάθος αξιολόγηση. Στο CCI τέλος, τα έσοδα είναι συνήθως αρκετά χαμηλά. Αναφέρεται αυτό στην έκθεση. Χρειαζόμαστε βέβαια προς την κατεύθυνση αυτή όχι μόνο ένα δίκαιο μηχανισμό για τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά και μια σφαγίδα ποιότητα, αν θέλετε, για τι επιχειρήσει που απασχολούν πολλού υπαλλήλου. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό ο κλάδο με τέτοιο υψηλό ποσοστό δημιουργικότητα να μαστίζεται από χαμηλόμιστες θέσεις από αβεβαιότητα, ανασφάλεια, γιατί προφανώ δεν θα έχουν και οι νέοι όρεξη στην περίπτωση αυτή να αναζητήσουν την τύχη του στον κλάδο αυτό. Αυτό θα θέλαμε να το αποφύγουμε. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και πάλι του εισηγητές γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή τους. Ε, e ε, Ευχαριστώ πολύ. μέλος και των δύο επιτροπών. Είμαι υπέρ της βιοτεχνικής δραστηριότητας γενικά και γι' αυτό είμαι υπέρ της εξιοποίησης ε, των βιοτεχνικών ικανοτήτων των ευρωπαϊκών λαών. Κατέθεσα και πρόταση ψηφίσματος. Στη Γαλλία η βιοτεχνία απασχολεί 3 εκατομμύρια 500 δραστηριότητες και επιτρέπει 100.000 προσλήψεις κατέτος. Δεν μετακινούνται αυτές οι δραστηριότητες και ε, βοηθούν το να διασωθούν οι διαγενειακές ε, ικανότητες, ε, τέχνες και ταλέντα. Καταπολεμάται η πειρατεία και η παραποίηση αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην θίξουμε τις εθνικές αρμοδιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και να μην αγνοήσουμε τις παραδοσιακές μορφές μαθητείας. Σχετικά με ένα κοινό ορισμό που θα διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Υπάρχει ο κίνδυνος να θέσουμε σε κίνδυνο τους ορισμούς που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να προστατεύσουν και να αξιοποιήσουν τις επιχειρήσεις. Όταν μιλάμε για θέματα επίσης χρηματοδότησης, αναφέρεστε στην δυνατότητα που παρέχει ο μηχανισμός εγγυήσεων και του Creative Europe. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα αποτελέσματα υπέρ των μικρομεσαίων δεν είναι εδώ. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων ποσών. Θα είμαι ιδιαίτερος παρούσα λοιπόν στα θέματα αυτά για να προωθήσουμε και να ακτινοβολήσουμε την πολιτιστική μας εξαίρεση. Ευχαριστώ συνάδελφε, αυτός ήταν ο πρώτος γύρος, τελείωσε. Θα δώσω τώρα την προεδρία στον συνάδελφο Ρούμπιχ για τον δεύτερο γύρο. Να ευχαριστήσω την Πρόεδρο Κώστα και για τις εισήγησει εισηγήσεις των ε, εισηγητών και των σκιωτών και τώρα θα θέλαμε να πράσουμε στο τμήμα όπου μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη. Δύο λεπτά κατά το όριο. Και έχουν ζητήσει κάποιοι ήδη το λόγο. Η κυρία Κάμερφερτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τους συζητητές. Νομίζω ότι είναι καλό σημείο κίνηση σε αυτό το οποίο έχουμε ενώπιον μας για τις περαιτέρω εργασίες μας και συζητήσεις μας. Και ελπίζω δε ότι στην τελική ανάλυση θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια καλή έκθεση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα και μόνο σημείο, για το οποίο πάντα πραγματικά με πιάνει μια κάποια νευρικότητα όταν το διαβάζω, το σημείο 8 της έκθεσης, όπου μιλάμε για τις πιο αυστηρές κυρώσεις σε ό,τι αφορά την εγκυμένη ανιχνευσιμότητα ως τρόπος αντιμετώπισης της πειρατείας. Εδώ μιλάμε για, το, για τα περιεχόμενα online. Και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι είμαι επί της αρχής κατά οποιασδήποτε παρακολούθησης και ανίχνευσης ψηφιακή επικοινωνία, γιατί είμαι υπέρ τη ελευθερία επικοινωνία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και να βρούμε άλλου τρόπου για την καταπολέμηση τη πειρατεία. Όταν μαθαίνουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία οι υπηρεσίε οι οποίε παρέχονται με ε, παράνομο τρόπο στο διαδίκτυο, μπορούμε να ακολουθούμε την προφανή λύση της διαγραφή των στοιχείων αυτών στην ε, Γερμανία το τελευταίο χρόνο είχαμε μία μεγάλη υπόθεση ε, και μπορούμε να πούμε ότι πλέον υπάρχει ένα ολόκληρο κλάδο δικηγόρων που ασχολείται μόνο με την αποστολή επιστολών ε, προειδοποιητηρίων προ του ε, καταναλωτέ. Ε, και φαίνεται, είναι πολλά υποσχόμενα τα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι όλα αυτά βοηθούν και στην, στον κλάδο της μουσικής. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε ως μέθοδο όχι τόσο τα θέματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και παρακολούθησης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Ρούμπιχ. Ο κύριος Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Co mnie najbardziej ucieszyło w tym sprawozdaniu? Po pierwsze, podkreślenie roli długofalowej polityki. Αυτό που μου στην έκθεση αυτή είναι το των μακροπρόθεσμων πολιτικών. Κατά δεύτερον, η ανάγκη προστασίας των δημιουργικών κλάδων με συνεκτικό τρόπο η καλύτερη ποιότητα υποβολής εκθέσεων και η καλύτερη αμοιβή των όσων απασχολούνται στις ε, βιομηχανίες αυτές, στον κλάδο αυτό. Και τέλος, θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τι με ανησυχείς όμως. Ε? Καταρχάς, ε, τα, η αξιοπιστία των στατιστικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε. Σε κάποιες περιπτώσεις ακούμε 3%, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ακούμε 15% σε ό,τι αφορά δηλαδή το ποσοστό του ευρωπαϊκού προπολογισμού που δαπανάται στην δημιουργική, στο δημιουργικό κλάδο. Γιατί, γιατί κανείς ε, δεν έχει κοινού ορισμούς, κοινού όρους ε, των δαπανών για τα θέματα τέτοια πολιτισμού και σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι σαφές το τι θεωρείται πολιτισμικό και τι όχι σε κάποια χώρα και φυσικά πολλές φορές υπάρχουν και διαφορές. Ένα πρόγραμμα για παράδειγμα μαγειρική στην τηλεόραση. Κάποιοι το αποκαλούν πολιτισμικό, κάποιοι όλοι, κάποιοι άλλοι όχι. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα συντονισμό όμω. Κατά δεύτερον, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο εξοδεύει χρήματα στι βιομηχανίε αυτέ. Καταρχάς είναι μονομένοι χρήστες που αγοράζουν διάφορα πράγματα. Και αυτοί χρηματοδοτούν τη δημιουργική βιομηχανία. Αυτή είναι η πρώτη. Κατά δεύτερον, οι επιχειρήσεις και μόνο στην τρίτη θέση. Βλέπουμε τις κυβερνήσεις. Θα πρέπει αυτό να το προωθήσουμε ως επιχειρήσμα, γιατί η αξιοπιστή των δύο επιτροπών μας εξαρτάται από την αξιοπιστία των δεδομένων που χρησιμοποιούμε. Τέλος, να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ήτρε. Γιατί στην Επιτροπή Πολιτισμού ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Η συμβολή λοιπόν της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας είναι πάρα πολύ σημαντική και ακόμα καλύτερα θα ήταν να υπήρχαν και εξέταση από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Τότε ενδεχομένως να είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και κάποιες αλλαγές και για την δημοσιονομική πολιτική και δημοσιονομικέ ρυθμίσει, γιατί και αυτέ είναι σημαντικέ για το μέλλον της ε, δημιουργικού κλάδου. Σα ευχαριστώ πάντως για του δύο εισηγητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος και η κυρία Τρούπολη επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μικρό ιστορικό. Η συζήτηση για αυτού του είδους τις οικονομικές δραστηριότητες ξεκίνησε πριν 15-20 χρόνια. Υπήρξε ένα βιβλίο ενός Αμερικανού συγγραφέα του Richard Freund που έλεγε, λεγόταν The Creative Class, η δημιουργική τάξη. Βασιζόταν στην γνώση, στον σεβασμό και στην ανοχή ιδιαίτερα απέναντι στους ομοφιλόφιλους. Ε, δεν είναι κάτι το αυστηρά οικονομικό, είναι κάτι το οποίο αφορά στο άνοιγμα της κοινωνίας σε αξίες όπως η ανοχή αλλά και τεχνολογία κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή πρέπει να είναι η λογική μας όταν συζητάμε τέτοιου είδους εκθέσεις για τις δημιουργικές αυτές οικονομικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες δεν αντικαθιστούν τις πολιτιστικές πολιτικές. Ε, ε, περιλαμβάνουν πολιτιστικά στοιχεία, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τμήματα της σύγχρονης, μιας σύγχρονης οικονομικής πολιτικής και πάνω σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε. Υπάρχει λοιπόν ένα συνδυασμός οικονομικών και πολιτιστικών πολιτικών, αλλά πέρα από αυτά τα οποία ακούστηκαν, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να έχουμε τα απαιτούμενα μέσα και τα απαιτούμενα προγράμματα για να στηρίξουμε τις δημιουργικές αυτές δραστηριότητες πέρα από το πρόγραμμα Creative Europe και χρειαζόμαστε και άλλα προγράμματα έτσι ώστε να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο τις δημιουργικές αυτές ε, οικονομικές δραστηριότητες. Όχι εις βάρος του Creative Europe, αλλά για να διευκρινίσουμε ότι αν θέλουμε πράγματι να είμαστε πιο επιτυχείς σε οικονομικό επίπεδο και στα πλαίσια των ΕΦΣΥ και στα πλαίσια των άλλων προγραμμάτων, χρειάζεται δυνατότητα στήριξης καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είμαι πεπισμένη ότι απαιτείται να υπάρχει μια πραγματική βιομηχανική πολιτική για την στήριξη αυτής της ε, πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας εισαγωγικά. Στην περίπτωση της παγκοσμιοποίησης είμαι βέβαιος ε, θα πρέπει σε επίπεδο διακανονιστικό να δημιουργήσουμε ένα πιο δυναμικό και προσαρμοστικό πλαίσιο είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί από εσά έχουν ήδη αναφερθεί στην προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωση στον τομέα της δημιουργικότητας, της βιοτεχνίας. Αναφερθήκατε στην ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Υπόθηκε και συμφωνώ μαζί σας ότι πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες δεν μετακινούνται τις περισσότερες φορές είναι κάτι λοιπόν το πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να στηρίξουμε και άλλωστε τα έσοδα από τον ψηφιακό τομέα είναι χαρακτηριστικά υψηλά και το 90% των ψηφιακών δεδομένων που υπάρχουν στον κόσμο έχουν, ε, είναι αντικείμενο παραγωγής τα τελευταία δύο χρόνια. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να υποστηριχθούν αυτές οι βιομηχανικές δραστηριότητες. Για την παραποίηση δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταπολεμηθεί, πρέπει να προστατευτεί η πνευματική ιδιοκτησία. Ξέρω ότι στη δική μου χώρα υπάρχουν κανόνες και νόμοι μετά από δύο προειδοποιήσεις μια ε, σύνδεση διαδικτυακή μπορεί πλέον να απαγορευτεί. Αλλά γενικά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να αναζητήσουμε τις πιθανές κυρώσεις που θα προστατέψουν τις δραστηριότητες αυτές που δημιουργούν θέσεις εργασίας και είναι βασικό. Ευχαριστώ. Μαραγάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Vamos a Θα πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο την έννοια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα μέσα. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν εσωτερικές αντιθέσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αναφέρουμε δύο θέματα, το οποίο έχει ήδη τεθεί. Σχετικά με τον πολιτισμό, οι δημόσιες επενδύσεις, τα δημόσια χρήματα, θα ε, πρέπει να πω ότι η κρίση των τελευταίων σχεδόν 10 ετών, σχεδόν 19 ετών, έχει λειτουργήσει καταστροφικά στις δημόσιες πολιτικές υπέρ του πολιτισμού σε κάποιες χώρες ε, περισσότερο από ό,τι σε άλλες, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου. Είναι εντυπωσιακή η αριθμή. Σύμφωνα με στατιστικές που προέρχονται, στατιστικές που προέρχονται από την Eurostat, το 2014 έχει πέσει πάρα πολύ το ποσοστό των χρημάτων που διατίθενται για πολιτιστικές δραστηριότητες. O en la Europa Central, en cambio, tenemos 148 euros por habitante en Alemania, 249 en Francia. Y en los países... Εν πάση περιπτώσει έχουν υπάρξει μειώσει ακόμα και στη Φιλανδία στον προπολογισμό για τι δημόσιε επενδύσει στον πολιτισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες και γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Θα πρέπει να οδηγεί σε σύγκληση και σε αύξηση των αριθμών αυτών και σε σενάρι πραγματικής ανάπτυξης και σύγκλησης. Υπάρχει επίσης και ένα γεωγραφικό blocking και ένας γεωγραφικός αποκλεισμός και σε επίπεδο πολιτιστικών προϊόντων και όχι μόνο τεχνολογίας, γλωσσικής, υπάρχουν ε, και καλυμμένοι θεμητοί ίσως εθνικοί προστατευτικοί κανόνες ε, και για την αγορά εργασίας και για τις βιοτεχνίες κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει επίσης να είναι ένας προσανατολισμός ως σαφής της έκθεσης αυτής. Εν πάση μετά από όλα αυτά θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές γιατί μας δημιούργησαν ένα εξαιρετικό πλαίσιο συζήτησης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συζητητές στο σημείο αυτό, γιατί το θέμα αυτό το επεξεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά μεταξύ των δύο συναρμοδίων επιτροπών και νομίζω ότι τελικά έχουμε μια πολύ καλή βάση ενώπιον μας. Ένα σημαντικό θέμα είναι η έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση μακροπρόθεσμου προγράμματος, ειδικά για την ε, δημιουργικό κλάδο, γιατί μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν είναι αμυγός οικονομικά ή αμυγός βιομηχανικά, αλλά έχουν και μια πολιτοσμική προστιθέμενη αξία. Πρόκειται για τις δύο πτύχες του ίδιου νομίσματος. Πάντα λοιπόν ε, θέτουμε και τις ε, διαστάσεις της κοινωνικές ε, και τις οικονομικές. Ε. Πρέπει για τα πράγματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς λοιπόν αυτή η πολυμορφία στην Ευρώπη είναι αυτή που είναι τόσο γόνιμη. Και αντίστοιχα θα πρέπει να απτυχθεί λοιπόν και ένα πλαίσιο πολιτικής. Κάτι άλλο το οποίο το λέμε εδώ και καιρό σε ό,τι αφορά τον πολιτισμικό κλάδο. Συχνά κοιτούσαμε μόνο τον πολιτισμικό κλάδο, αλλά δεν είναι λαμβανόταν υπόψη είναι ο πολιτισμικός κλάδος ή ο οικονομικός κλάδος. Και σε ό,τι αφορά λοιπόν την περιγραφή των ε, προγραμμάτων θα πρέπει να θέσουμε σημεία επικέντρωσης και σημεία προτεραιότητας. Γιατί συχνά υπάρχει μια σύνδεση με μια συγκεκριμένη περιοχή, όπου δεν μπορεί να υπάρχει και εξωτερική ανάθεση. Θα πρέπει λοιπόν, όπως είπε και ο εισηγητής, να υπάρχει μια προώθηση ε, τοπικών ε, πρωτοτύπων επιχειρήσεων και επαγγελμάτων. Και νομίζω ότι μπορούν να υποστηριχθούν αυτά με μεγαλύτερη χρηματοδότηση και θα πρέπει να κάνουμε και τι συζητήσει αυτέ αν θέλετε, με διαφορετικό τρόπο σε ό,τι αφορά την παροχή διαφορετικών οικονομικών πλαισίων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ε, ε, κλάδο τη δημιουργικότητα και τον κλάδο των ε, πολιτισμικών. Προσβλέπω λοιπόν στην καλή συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε το δυναμικό για κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει πριν από πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ, ο δεν βλέπω να ζητά κανεί άλλο το λόγο. Και έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε και θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο για να τοποθετηθεί. Έχουμε τον προϊστάμενο της σχετικής γενικής διεύθυνσης και θα ήθελα να κάνετε μια δήλωση δύο-τρία λεπτά παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω και την κυρία Κώστα, την πρόεδρο. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη αυτή η έκθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ και την ε, προσοχή που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία. Νομίζω ότι οι συγητές ανέφεραν ότι υπάρχει ένα αναδυόμενο πλαίσιο, το οποίο όμως δεν έχει αναδυθεί ακόμα. Υπάρχουν ε, εργασίες εν εξελίξη, οι οποίες θα συνεισφέρουν ιδιαίτερο σε αυτό το πλαίσιο. Να σας υπενθυμίσω τι κάνουμε για την ψηφιακή ενέα αγορά. Όπως γνωρίζετε υπάρχει μια αναθεώρηση για τα πνευματικά δικαιώματα που είναι πρώτων πυλών, ολοκληρώνεται ε, μάλλον το Σεπτέμβριο και θα εξετάσει κάποια από τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα, ε, συμπεριλαμβανομένες και της δίκαιης αποζημίωσης των δημιουργούν και το λεγόμενο κενό χάσμα αξίας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά ε, και το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν τόσο μεγάλο ε, κατανάλωση πολιτιστικού περιεχομένου ενώ ταυτόχρονα είναι τόσο μικρές οι αμοιβέ ε, για τους δημιουργούς. Επίσης θα δούμε την αξιολόγηση για την αμοιβή των ε, δημιουργών και την κατάλληλη ε, χρηματοδότηση της δημιουργικής διαμηχανίας. Επίσης υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία. Θυμάμαι ότι έγινε μία παρουσίαση ε, στην Επιτροπή Πολιτισμού από τη Eurostat που έδειξε τι ακριβώς κάνουμε. Η δουλειά αυτή απαιτεί χρόνο, διότι όπως είπαμε υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί, δεν συλλέγουν όλα τα κράτη-μέλη δεδομένα με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει αυτή η δουλειά, διότι σε αντίθεση με τις μελέτες είναι εργασίες οι οποίες συνεχίζουμε κάθε χρόνο και έχουμε καλά αποτελέσματα, διότι τα κράτη-μέλη χωρί να τους επιβληθεί κάποιος ορισμός ε, τείνουν να συγκλίνουν και επομένω, ε, είναι πολύ σημαντικό να ε, υποστηρίξουμε αυτή τη δουλειά. Να σας πω τι κάνουμε με τις περιφέρειες, διότι κάποιο ανέφερε ότι, στην έκθεση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο των περιφερειών για την ε, καθορισμό των στρατηγικών. Τουλάχιστον 7 περιφέρειες έχουν θεωρήσει τον ε, ε πολιτισμό και τη δημιουργία ως σημαντικού τομεί στις πλατφόρμες που θέλουν να δημιουργήσουν. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για το συντονισμό, για πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μέτρα ε, καινοτομία. Υπάρχουν κάποια πιλωτικά προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν από τη Δημιουργική Ευρώπη. Έχουμε περιορισμένους μεν πόρους, αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κόμβους, μία πλατφόρμα για δημιουργικούς επιχειρηματίες, ε, επιχειρηματίες δηλαδή του κλάδου της δημιουργίας, ε, και γι' αυτό ακριβώ και περιμένουμε με ανυπομονησία την έκθεσή σα. Αν μπορώ να τα συνοψίσω, συμφωνούμε με την ανάλυση, υποστηρίζουμε τη φιλοδοξία, περιμένουμε με ανυπομονησία την έκθεση και είμαστε στη διάθεσή σα για οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε να σα παράσχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρατε γιατί το θέμα δηλαδή είναι όταν ε, αγοράζει κανεί μια συσκευή και τη χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, σήμερα, πρέπει να αποδεχτεί τι γενικότερε συνθήκε ε, που ισχύουν. Και παρόμοια υπάρχουν όρια για την πρόσβαση σε τέτοια περιεχόμενα. Υπάρχουν κάποιοι γενικοί όροι χρήση. Θα πρέπει αυτό να ρυθμιστεί ε, αντίστοιχα όπω ε, και στα άλλα προϊόντα σε ό,τι αφορά τις άντρε και ό,τι αφορά του καθεξής. Αυτό θα έχει μεγάλη επιρροή και να μιλήσουμε και με, την, με τον Κάλο Κουράτσα από την Γενική Διεύθυνση Κρός. Oui, merci beaucoup. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και θα συμφωνήσω εγώ με τα σχόλια του κυρίου Τζαμπιέρη. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί πλήρως πόσο σημαντική είναι η οικονομική ε, δραστηριότητα για τις θέσεις εργασίας στον τομέα αυτών και όπως ε, ακούσατε θα δημοσιεύσουμε μια έκθεση που επισημαίνει τη σημασία αυτού του κλάδου. Επίσης, ε, σημειώνουμε και την άποψη των επιτροπών ε, του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο σωστή και πιο συνεκτική πολιτική. Είμαστε ήδη, όπως σας είπε ο συνάδελφος Τζαμπιέρη, ε, καθοδόν για να υλοποιήσουμε διάφορες ε, δράσεις και στο κόσμο και στον ορίζοντα 2020. Ο κύριος Τζαμπιέρη σας επεσήμανε τη σημασία της ε, στρατηγικές ε, και της συνεργασία με τις περιφέρειες για την ευφυή e e, εξειδίκευση. Συνεργαζόμαστε με τις ε, η Επίτροπος Μιανκόφσκα είπε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ε, ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε για να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ τουρισμού και πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι ένα πιο συνεκτικό πλάσιο μπορεί να απαιτείται σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό και ε, βλέπουμε πολύ ευνοϊκά τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Μοργάνο, τον εισηγητή μας, για μια σύνοψη και ενδεχομένω ε, μια ερμηνεία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ διότι είχαμε 13 διαδοχικές παρεμβάσεις ε, και πολλά στοιχεία επί της ουσίας και αυτό βοηθούν ιδιαίτερα τη δική μας δραστηριότητα και κυρίως ε, το γεγονός ότι συμμερίζονται τις απόψεις μας και οι δύο παρεμβάσεις που ακούσαμε προηγουμένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι πολύ σημαντικά. Τι να προσθέσω εγώ για τα πολλά αιτήματα με τα οποία συμφωνούμε σε γενικές γραμμές και δεν ε, πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια έκθεση η οποία θα είναι πλήρης ευθύς εξ αρχής. Ε, θέλαμε με τη συνεισφορά των συναδέλφων να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την πρόταση αφού θα δώσουμε εμείς κάποιες πρώτες κατευθύνσεις. Καταρχάς, κατά την άποψή μας είναι ε, πιο σημαντικό να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Ποιος είναι ο φαύλος κύκλος? Η υποτίμηση του κλάδου. Το γεγονός ότι υπάρχει ε, ισχνό ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν αιτήματα από την αγορά εργασίας χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη προσφορά εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο ε, το οποίο ε, διέπει τη λογική μας. Τώρα, όσον αφορά τις ε, προϋποθέσεις υλοποίησης. Επιμένω διότι η προσπάθεια που κάνουμε δεν είναι να παρουσιάσουμε μια ωραία έκθεση και να σταματήσουμε εκεί, αλλά θα θέλαμε να περάσουμε από την έκθεση σε μια συνεχή δέσμευση όπου φυσικά και οποιαδήποτε απόπειρα για να έχουμε ένα πιθανό ορισμό του κλάδου θα μας βοηθήσει ώστε η έλλειψη ορισμού να μην επιτρέπει και την έλλειψη χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ακριβώς αναφερθήκαμε και στα στοιχεία. Το γεγονός ότι πρέπει να συλλέγονται στοιχεία από κάποια δομή όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Κοράτσα, αλλά και ο ορισμός των στατιστικών, ε, κυρίως στο σημείο 3 που αναφερόμαστε σε στατιστικούς ορισμούς για να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια, γιατί αλλιώς είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τα στοιχεία. Και πρέπει επίσης να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι καθοριστική σημασία σήμερα. Αν όντω ε, ισχύει ότι το 90% που ισχύει είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτό. Επομένως, ε, το πώς μπορεί κάποιος να εξαρχηριώσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για να μπορέσει να υπάρχει κατάλληλη αμοιβή, γιατί αλλιώ υπάρχει μια αντίφαση. Απ' τη μια υπάρχει μια πολύ σημαντική όθηση και ε, όταν πρέπει κάποιο να λάβει πόρους για να αναπτυχθεί, σταματάμε και πρέπει λοιπόν να βρούμε και έναν τρόπο ώστε να προχωρήσει και το ζήτημα αυτό. Είναι σαφές ότι δεν είναι εύκολο αυτό, διότι σήμερα στον τομέα της ψηφιοποίησης υπάρχει ένας τομέας ο οποίος πράγματι χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες ε, διατάξεις οι οποίες συζητώνται αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στα όσα υπενθύμησαν και κάποιες παρεμβάσεις. Κάποια κοινωνική Στάτου ε, στάτους των ε, δημιουργών, κάποια αναγνώριση. Υπάρχει και ένα έγγραφο του 2007 το οποίο ήδη αναφερόταν στο θέμα αυτό, επομένως πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και στο θέμα αυτό και για λόγους ομοιομορφίας, να λάβουμε υπόψη τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα μεταξύ των 27 πλέον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως για τη συνεισφορά σας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ ε, και για τις τροπολογίες και για τις ε, προτροπές που θα έχουμε και τις παρατηρήσεις. Λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που μας είπατε και θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τη δουλειά μας τις επόμενες ημέρες. Θα ήθελα να στραφούμε λίγο προς το μέλλον. και όχι εξ ονόματος της Ήτρε, αλλά γενικά θα ήθελα να διευκρινίσουμε λίγο τις θέσεις σας. Ίσως να είμαστε λίγο, θα έλεγα, έντονοι. Δεν πρέπει να φανούμε υποχωρητικοί όμως. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ε, διευκολυντικά για τα οικονομικά συμφέροντα αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρχουν τέτοιου είδους οικονομικές δραστηριότητες στην Ευρώπη χωρίς τον πολιτισμό. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα ευρύτερα. Το θέμα είναι ότι έχει ενταχθεί στο FC, όχι γιατί το θέλει η Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά γιατί εμείς το βάλαμε. για το θέμα των αμοιβών. Αναζητώντας συμμαχίες, ο τομέας αυτός φαίνεται λίγο τοξικός θα έλεγα. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα λιμάνι προστασίας, σωτηρίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες της άνησης σχέσης δημιουργών και ε, με τις πλατφόρμες οι οποίες μεταφέρουν το έργο τους. η βιομηχανία, ηλιανική ας πούμε μάλλον οικονομική δραστηριότητα σε μια άλλη πλευρά του κόσμου είναι αυτή η οποία αποφασίζει για το πόσο θα αμείβεται η αγορά ή η παραγωγή του χάλιβα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Συνεπώς λοιπόν αν συνδυάσουμε την δημιουργική δραστηριότητα των δημιουργών ακριβώς, των καλλιτεχνών με οικονομικά κριτήρια ε, σε μια πλατφόρμα ευρύτερη και εφόσον η πλατφόρμα σέβεται γενικά τα δικαιώματα και τους κανόνες, αλλά αυτό δεν ισχύει βέβαια. Μιλάμε για μια οικονομική δραστηριότητα και δεν θα δεχόμαστε παράνομες δραστηριότητες γύρω από αυτήν σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, πόσο μάλλον στον πολιτισμό. Μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο μόχλευσης, όχι ίσως όπως γίνεται σε άλλους τομείς, αλλά δεν πρέπει να αγνοηθεί. Τώρα για τα πιο επιμέρους οικονομικά θέματα έχει δημιουργηθεί μερικές φορές για τους δημιουργούς μια δύσκολη αν θέλετε κατάσταση. Όταν μιλάμε για άειλα προϊόντα, άειλα αγαθά, είναι πολύ δύσκολο να τα εντάξει κανείς σε ένα απολογισμό οικονομικό. Ο τομέας αυτός βρίσκεται σε μια πιο προβληματική κατάσταση από ό,τι στο παρελθόν. Οι μικροπιστώσεις είναι προβληματικές δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολύ μικρών μονάδων ε, και η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι στο παρελθόν επαναλαμβάνω. Αν το δούμε σαν τομέα και όχι σαν κάτι το αφηρημένα πολιτιστικό, θα υπάρξει μια σωστότερη αντιμετώπιση σε επίπεδο μιας σεβαστής οικονομικής δραστηριότητας. Και έτσι δεν θα εξαιρούνται οι δραστηριότητες αυτές ε, από την χρηματοδότηση. Δεν ισχύει αυτό για άλλους τομείς. Με την ίδια λογική θα έπρεπε η αεροναυτική σαν παράδειγμα να μην χρηματοδοτείται γιατί πολλές φορές αναφέρεται σε κάτι το άειλο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κάπως έμονοι, πρέπει να είμαστε κάπως ισχυροί στον τρόπο με τον οποίο διεκδικούμε αλλά η ηθική υπεροχή του θύματος μπορεί να εντυπωσιάζει, αλλά δεν μας οδηγεί και πουθενά. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε μια σωστή εταιρική σχέση και να διασφαλίσουμε τη σωστή μόχλευση για το ευρωπαϊκό μέλλον. Ο πολιτισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού μέλλοντος, έχει σχέση και με την παγκοσμιοποίηση, ε, έχει σχέση με έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους τομεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα στους δύο εισήγητες και τα μέλη του Κοινοβουλίου που συμμετείχαν σε όλη τη διαδικασία και όλους τους προσκεκλημένους. Είναι καλό να κάτσουμε να σκεφτούμε το θέμα αυτό λίγο κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Για την Ήτρε. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η έκτη Σεπτεμβρίου. Έχουμε χρόνο λοιπόν να κάνουμε βελτιώσεις. Επόμενη συνεδριάση στις 13 ε, Οκτωβρίου στην Ήτρα. Και η ψηφοφορία στην ε, Ήτρα θα λάβει χώρα στις 10 Νοεμβρίου σε κοινή συνεδρίαση την οποία θα διεξαγάγουμε από κοινού να σας ευχαριστήσω όλους και να παραδώσω εκ νέου τα ενία της Προεδρίας στη συνάδελφο Κώστα. Σας ευχαριστώ για την ε, πρώτη αυτή κοινή συνεδρίαση που θεωρώ ότι αποτέλεσε σημαντική επιτυχία. Και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ρούμπιχ. Ε, πιστεύω ότι πρόκειται για μια υπέροχη πρωτοβουλία. Καλά κάναμε και επιθυμήσαμε αυτή την ε, συνάντηση και τη συνεργασία θα επαγρυπνούμε για αυτή την πολύ σημαντική γνωμοδότηση, έκθεση συγγνώμη, και για μένα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τρει επισημάνσει. Η συνάδελφο Ζρογεύσκη αναφέρθηκε στο θέμα των δεδομένων. Πιστεύω ότι υπάρχει μια σχέση, ε, μια έρευνα ε, στην οποία αναφέρεται, ε, διότι ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι το θέμα των δεδομένων για δύο λόγους. Δεν έχουν όλα τα ίδια μέλη τα ίδια κριτήρια, αλλάζει η παράμετρος ανάλογα με τις αναλύσεις και επομένως ε, ε, τελικά έχουμε διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία. Καλό θα ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε από μεθοδολογική σκοπιά κάτι για τα ε, δεδομένα και καλό θα ήταν να το αναφέρετε στην, στην έκθεσή σας. Δεύτερον, εδώ βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εν γένει ο πολιτισμό, και γι' αυτό λυπούμαστε, πρέπει να αποδείξει πάντα κάτι για να θεωρηθεί ο σημαντικό. Επομένως, ε, ε, αναρωτιέται κανείς ποια είναι η οικονομική αξία του πολιτισμού. Η, ε, ε, ο πολιτισμός έχει μια αξία αυτός καθεαυτός και από εκεί και πέρα υπάρχει και η οικονομική του αξία αντιληφθήκαμε ότι χωρίς δημιουργικότητα, χωρίς πολιτισμό, χωρίς δημιουργός, χωρίς ταλέντα δεν υπάρχει ε, βιομηχανική πολιτική. Αυτό είναι ήδη ένα θέμα το οποίο από μόνο του θα δικαιολογούσε αυτή την έκθεση γιατί δεν ήταν πολύ εύκολο ο διάλογος και μεταξύ των επιτροπών μας και εγώ είμαι περήφανη που συνεισέφερα ως πρόεδρος μαζί με τον συνάδελφο Μπούσεκ και τον κύριο Ρούμπιχ ε, ώστε να προχωρήσει αυτή η συνάντηση διότι πρέπει να γίνει και σε επίπεδο επιτροπή. Είναι πολύ καλό βλέπουμε ότι οι τμήματάρχες συνεργάζονται και υπάρχουν διάφορα τμήματα τα οποία συνεργάζονται όταν δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να συνεργάζονται. Ε, συγγνώμη, αλλά είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι μόνο θέμα μεθόδου, αλλά θέμα ισίας. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, η χρηματοδότηση που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι, υπό την έννοια ότι όπως έλεγε από τη μία και ο κύριος Έλλερ και ο κύριος Μόργανο, έχουμε θέμα ιδιωτερότητα του συγκεκριμένου κλάδου στην Δημιουργική αύριο και αύριο, Ευρώπη και αύριο θα παρουσιάσουμε την πρώτη ε, εκτελεστική έκθεση ε, υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι επιτέλους αύριο θα το δούμε, ε, υπήρξε και συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Υπάρχει ένα νέο ταμείο το οποίο δεν έχει τεράστια κονδύλια αλλά είναι εγγύηση ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα απευθύνεται ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα το οποίο ε, θεωρητικά δεν έχει πρόσβαση σε αυτή τη ε, δανειοδότηση. Ε, και εμείς είμαστε πιο φιλόδοξοι, το συζήτησα και με τη Γενική Διεύθυνση Connect και πέραν της ΕΑΚ. Ακούω συνέχεια ένα θόρυβο, κάντε μου λίγο τη χάρη. Πρέπει λοιπόν οι πόροι του Ταμείου να συνδυαστούν με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, διότι πρέπει να υποχρεώσουμε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να υπάρχει μια αναφορά, διότι δεν υπήρχε η αναφορά στις προτεραιότητες και στη δημιουργική βιομηχανία. Θέλουμε να έχουμε μια συνεκτική πολιτική που να αφορά και αυτά. Εγώ μίλησα και με τη Γενική Διεύθυνση Connect και είπα ότι κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να περιμένουμε να έρθουν τα προγράμματα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκές πλατφόρμες για τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία και σας το λέω διότι ήδη το συζητάμε εμείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήμουν πιο φιλόδοξη, θα το συζητήσουμε αύριο και θεωρώ ότι όπως έλεγε και η συνάδελφος Τρούπελ και το λέω αυτό μόνο για αυτά που θα πω αύριο ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία, αλλά χάθηκε λίγο στον τομέα της ε, δημιουργική και πολιτιστικής βιομηχανία, διότι δεν έγινε το πρόγραμμα της εγχώνευσης και έχουμε τώρα τον πολιτισμό που δίνει πολύ μεγαλύτερη ε, ε, σημασία στα μη κερδοσκοπικά στοιχεία παρά το γεγονός ότι έχουμε πλέον ε, και κερδοσκοπικά. μετά έχουμε το ακουστικά. Και πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα νέο έξονα που θα πρέπει να είναι η δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία. Τα λέω αυτά προλαμβάνοντας λίγο τα αυριανά, αλλά πρέπει να είμαστε εξαφείς ως προς τη φιλοδοξία που πρέπει να έχουμε. Για να ολοκληρώσω, ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα των αμοιβών των καλλιτεχνών και επίσης ε, ε καταπολέμωση της, μορφ... της πειρατείας, διότι είναι και μεγάλη φορολογική ζημία. Δεν είναι μόνο ζημία στον πολιτισμό και φυσικά υπάρχει και ένα θέμα το οποίο αφορά κάτι το οποίο θα σας φανεί μακρινό, αλλά είναι πολύ σημαντικό και θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον για αυτή τη νέα προσήκηση. Η δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία θα πρέπει να έχει ε, κάποιο χώρο και στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμικής Κληρονομιάς, το οποίο επιτύχαμε για το 2018, θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, της Επιτροπής Ήτρα, ξεκινώντας από τον Επίτροπο Ρούμπιχ, να μας υποστηρίξουν, διότι διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ ε, για το 2017 και το έτος είναι για το 2018. Δεν γνωρίζουν καν το πρόγραμμα, ζητήσαμε ε, να έχουμε το πρόγραμμα το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να κάνουμε από κοινού αυτή τη μάχη και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε πολλά στοιχεία και για τον πολιτισμό. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τον πρόεδρο Ρούμπιχ, τους συναδέλφου από την Επιτροπή Πολιτισμού και την Επιτροπή Βιομηχανίας, να ευχαριστήσω τις δύο γραμματείες που ε, συνεισέφεραν ιδιαίτερα και υπήρχε μια συνεργασία που δεν ήταν δεδομένη και η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνεί που άντεξαν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ.